λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, είναι μεγάλη τιμή και ευχαρίστηση για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Μετά από δέκα έντονες μέρες όπου η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία απέδειξε την αριστεία της. Εφόσον επιβεβαιωθώ θα είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δημιουργήθηκε και γεννήθηκε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πνεύμα συνεργασίας και πολιτικού διαλόγου. Το 2014 είναι ένα ειδικό, ένας ειδικός χρόνος για την Ευρώπη. Εκατό χρόνια πριν είχαμε την αρχή δύο αυτοκτονικών πολέμων. 70 χρόνια πριν είχαμε την αρχή της απελευθέρωσης της Δυτικής Ευρώπης στα πλαίσια αυτού που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση οι ομάδες των κρατών δεν αναζητούσαν την ασφάλεια και την ευημερία με την δύναμη και την κυριαρχία αλλά με την ειρήνη και την ασφάλεια. Χρειάστηκαν να περάσουν αρκετά χρόνια και μόνο πριν 25 χρόνια η ιδέα αυτή έγινε ε, προσιτή για όλους τους Ευρωπαίους. Όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου ε, σταμάτησε και η βία και η κυριαρχία που ε, είχαν γίνει η μάστιγα της Ανατολικής Ευρώπης. Ε, το Ανατολή και Δύση έγιναν όπως είχε πει ο Βάκλαβ Χάβελ αυστηρά γεωγραφικοί προσδιορισμοί και όχι πολιτικοί ή και ηθικοί δεοντολογικοί. Η μεγαλύτερη κόρη μου γεννήθηκε το 1986 όταν το τέλος της ε, ευρωπαϊκής διέρεσης ήταν κάτι που δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ο μεγαλύτερος γιος μου το 89 όταν το, αυτό που δεν πίστευε κανείς έγινε πραγματικότητα και ο νεότερος το 4 το 2004 όταν πλέον οι νέες 10 χώρες ε, είχαν ήδη ενταχθεί στην Ένωση. Έχει σημασία να δούμε πού βρισκόμασταν όταν βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα και μη με παρεξηγείτε τα προβλήματα είναι σοβαρά. Εάν επιβεβαιωθεί η Επιτροπή Γιούνκερ πρέπει να είναι σοβαρή στην αντιμετώπιση τους και αυτή. Δεν ξεκινάμε όμως τόσο άσχημα όσο λέγουν ορισμένοι αρκετά συχνά. Η Ευρώπη ήταν ικανή να αλλάξει τις κοινωνίες. Η Ευρώπη απέφυγε την πολυδιάσπαση και τους οικονομικούς και νομισματικούς πολέμους και αντιμετώπισε και ε, την καταστροφή την οποία πολλοί επέσιαν στα πλαίσια της χειρότερης κρίσης μετά το 1930. Ε, υπάρχουν προβλήματα βέβαια και τα μέτρα είναι οδυνηρά για πολλά εκατομμύρια Ευρωπαίων που δεν έχουν δουλειά και δεν έχουν πολλές ευκαιρίες. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές. Θα πρέπει σαν πολιτικοί εμείς ε, να διαβεβαιώσουμε τους εκλογείς μας ότι αξίζουμε να μας εμπιστεύονται και θα μπορέσουμε να τους ικανοποιήσουμε. Εφόσον μας επιβεβαιώσετε θα χρησιμοποιήσω όλη μου την ενέργεια και την εμπειρία για να υποστηρίξω τον υποψήφιο πρόεδρο Γιούνκερ έτσι ώστε να πετύχει ε, το πρόγραμμά του για απασχόληση, ανάπτυξη και δημοκρατική αλλαγή. Θα πρέπει να δείξουμε με πρακτικό τρόπο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και τα ευρωπαϊκά όργανα δεν είναι αυτοσκοπή αλλά εξυπηρετούν τους πολίτες και τα κράτη-μέλη. Αυτά που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα κάνει γιατί μόνο αυτή μπορεί να τα κάνει και τα υπόλοιπα θα τα κάνουν τα κράτη καλύτερα από αυτήν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να συγκεντρώσει την, επιτροπή, την ε, προσοχή της εκεί όπου μπορεί να βοηθήσει. Οι κατευθυντήριες πολιτικές γραμμές του κυρίου Γιούνκερ, του υποψηφίου Προέδρου της Επιτροπής, θα, θα υποστηριχθούν από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως επίσης και από τις στρατηγικές προσανατολιστικές γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου. Καλύτερες νομοθετικές ρυθμίσεις, σωστότερες και ισχυρότερες διοργανικές σχέσεις είναι σεβασμός επίσης του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγματα απαραίτητα για να αρχίσουν τα πράγματα να βελτιώνονται. Να δούμε ποιες είναι τώρα οι κοινέ πολιτικές μας προτεραιότητες. Εάν με επιβεβαιώσετε από τις αρχές του επομένου έτους θα προτείνω στο σύνολο των επιτρόπων κάποιες προτάσεις οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα και καιρό και θα πρέπει να αποσυρθούν αφού τις συζητήσουμε μαζί σας. Μέσα σε ένα χρόνο θα παρουσιάσω μια ε, ε, μια επισκόπηση θα έλεγα των ε, βελτιώσεων στον τομέα της νομοθεσίας για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τα συμφέροντα της Ευρώπης. Αν το πετύχουμε αυτό είμαι βέβαιος ότι θα γίνει μια σωστή πολιτική συζήτηση για τον πολιετή προγραμματισμό σύμφωνα με το άρθρο 17 της συνθήκης εφόσον μας επιβεβαιώσετε στη θέση αυτή. Θα βελτιώσουμε επίσης και το σύστημα αξιολόγησης των επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ενθαρρύνουμε το Συμβούλιο να ακολουθήσει την ηγετική θέση, την πρωτοπορία την οποία έχει επιδείξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σαφές ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει θα πρέπει να ληφθούν υπόψη βέβαια. Έχει μεγάλη σημασία και η Επιτροπή, ε, το Συμβούλιο μάλλον αξιολόγησης επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να δράσουν και να κρίνουν ανεξάρτητα. Εγώ θα εκφράζω την άποψή μου για τις εκθέσεις αυτές όταν παρουσιάζονται στην Επιτροπή και όταν χρησιμοποιείται μια κίτρινη ή πορτοκαλή κάρτα, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το αντιμετωπίζει πολύ προσεκτικά, θα πρέπει η Επίτροπη να είναι σε στενότερο διάλογο με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Εφόσον με εγκρίνεται, ρόλος μου θα είναι να ενθαρρύνω τους συναδέλφους μου να συζητούν άμεσα με τα κοινοβούλια των κρατών μελών και να ακούν τις απαντήσεις και τις ερωτήσεις και να δίδουν και απαντήσεις. Τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων θα πρέπει να τα μοιραζόμαστε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να καταλάβουμε όλοι πραγματικά τι σημαίνει επικουρικότητα, κάτι που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφύγει τις μη απαραίτητε προτάσεις, έτσι ώστε να υπάρχει βέλτιστη δυνατή παρέμβαση όπου αυτό είναι απαραίτητο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα εθνών και πολιτών πει τις τελευταίες δεκαετίες. Ήρθαν κοντά ο ένας τον άλλο χωρίς να αμφισβητήσουν ποτέ την εθνική τους ταυτότητα ή τη σημασία των κρατών εθνών. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι ισχυρή μόνο αν τα κράτη-μέλη είναι ισχυρά και η ισχύ ε, ε, των κρατών μελών εξαρτάται και από την ισχύ της Ένωσης. Η προσωπική μου εμπειρία μου λέγει ότι μόνο από κοινού θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε θέματα σφαιρικά όπως οι κλιματολογικές αλλαγές, η τρομοκρατία και να αντιμετωπίσουμε ε, με θετικό τρόπο τις επιλογές κυριαρχίας και ανεξαρτησίας χωρών όπως η Ουκρανία. Κράτη λοιπόν και πολίτες είναι τα βασικά συστατικά της Ένωσης. Θα αποτύχουμε αν δεν λάβουμε υπόψη μας και τα δύο αυτά στοιχεία. Είναι στη φύση των πολιτικών σωμάτων να δώσουν περισσότερη προσοχή σε νέες πρωτοβουλίες και στην αξιολόγηση της υπάρχουσας νομοθεσίας. Θα πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Απαιτείται να γίνουμε καλύτεροι ακούγοντας τους πολίτες μας και τις επιχειρήσεις οι οποίοι είναι αυτοί που εφαρμόζουν την νομοθεσία και θα πρέπει να είμαστε απολύτως βία ειλικρινείς θα έλεγα όταν περιγράφουμε το τι δεν πάει καλά και πρέπει να αλλάξει ή όπου έχουμε αποτύχει. Θα πρέπει λοιπόν οι εμπλεκόμενοι όχι απλά να τους συμβουλευόμεθα εδώ στις Βρυξέλλες αλλά να εκπροσωπούνται σωστά εδώ στις Βρυξέλλες. Απαιτείται μεγαλύτερη επίσης διαφάνεια. Γι' αυτό θα προωθήσω και μια διοργανική συμφωνία για ένα υποχρεωτικό κατάλογο των καταγεγραμμένων λόμπις. Ε, δεν μιλάμε για έλλειψη νομοθεσίας, ε, για απελευθέρωση στον τομέα το διακανονιστικό, όχι, μιλάμε για μείωση της γραφειοκρατίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις, να δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης ε, και να αποφεύγονται απαράδεκτες και μη χρήσιμες νομοθετικές ρυθμίσεις. Θα αποτύχει η προσπάθειά μας αν επιτίθεται στα κοινωνικά δικαιώματα και την περιβαλλοντική προστασία. Εάν πράγματι θέλουμε εμείς να γίνουμε καλύτεροι νομοθετικά, τότε θα έρθουμε σε στενότερη επαφή με τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι απογοητεύονται γιατί πιστεύουν ότι η Ευρώπη είναι η πηγή της γραφειοκρατίας. Εγώ δεν είδε ο σε σχέση με αυτό. Προσπαθώ να σκεφτώ πρακτικά και προσπαθώ προσπαθώ να είμαι και επιλεκτικός εκεί που χρειάζεται. Εφόσον με επιβεβαιώσετε στη θέση μου θα στηρίξω τους συναδέλφους μου ε, στις σωστές τους επιλογές και θα σημειώσω τη διαφωνία μου με τις μη σωστές επιλογές. Γιατί ο κόσμος μας βλέπει όλους σαν ένα πράγμα. Λένε ποιοι, α οι Βρυξέλλες, πηγή απογοήτευσης ανεξάρτητα από τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε κατηγορώντας τα άλλα κοινοτικά όργανα δεν είναι κάτι που βοηθάει. Εμείς θα πετύχουμε μόνο αν από κοινού πολεμήσουμε και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να αλλάξουμε. Γιατί αλλιώς ε, δεν ε, θα δείξουμε ότι καταλαβαίνουμε το πόσο κατεπίοντα είναι τα προβλήματα. Θα σεβαστούμε βέβαια τις ευρωπαϊκές αξίες και τις αρχές μας, αυτά που μας ενώνουν μέσα στη διαφορετικότητά μας. Θα είμαστε επίμονοι στην εφαρμογή του νόμου από τα ευρωπαϊκά όργανα και από όλα τα κράτη-μέλη. Αν αποτύχει ένας από εμά επηρεάζεται και θίγεται η αξιοπιστία όλων μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακας της συνθήκης και της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι υπεύθυνη για την σωστή εφαρμογή τους. Θα είναι προσωπική μου ευθύνη ε, το να δώσω ε, επίσης προτεραιότητα σε αυτήν την συγκεκριμένη αρμοδιότητα την τόσο σημαντική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαβεβαίωση λοιπόν του σεβασμού και της εφαρμογής του κράτους δικαίου και του νόμου μαζί με τους συναδέλφους στο σύνολό τους. Και όταν πάρουμε την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα πάρουμε τα απαιτούμενα βήματα έτσι ώστε να δούμε τι θα γίνει και σε σχέση με τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, θα συνεργαστώ με όλες τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις που έχουν σαν στόχο την προώθηση και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η επιτυχία του ενός είναι επιτυχία όλων, γιατί όλοι συμμεριζόμαστε, όλοι συμμεριζόμαστε έλεγα τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για μεγαλύτερη πολιτική εμπλοκή στον τομέα αυτό, όπως έχετε και εσείς υπογραμμίσει θα οργανώσω ένα ετήσιο συνέδριο για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη, με την πλήρη συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων, των σχετικών όπως και του Κοινοβουλίου προφανώς. Αγαπητά μέλη, κυρίες και κύριοι, εισαγωγικά σας μετέφερα κάποιες σκέψεις γιατί τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά εφόσον με επιβεβαιώσετε στη θέση αυτή. Θεμελιώδη δικαιώματα καλύτερη νομοθετική ρύθμιση και μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υπηρετεί τους Ευρωπαίους. Φυσικά ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός. Είμαι στη διάθεσή σας για να σας ακούσω, να δεχθώ τις ερωτήσεις σας και να ξεκινήσει ένας πραγματικός πολιτικός διάλογος. Αυτά που προτείνουμε δεν είναι εύκολα και δεν είναι κάτι το δεδομένο. Οι αλλαγές είναι δύσκολες. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε οργανωθεί η ε, μία αλλαγή όμως ε, θα είναι κάτι το πάρα πολύ πιο οδυνηρό. Η αλλαγή την οποία προτείνει η Επιτροπή Γιούνκερ είναι θεμελιώδης αν θέλουμε πράγματι να αναπτυχθεί και να ξανάρθει η ελπίδα στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να πετύχουμε δεν θέλουμε μόνο την στήριξή σας αλλά την πλήρη εμπλοκή σας. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και μερικές φορές μπορεί να απογοητευτούμε. Αλλά όμως μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι παππούδες μας και οι γονείς μας είναι ότι τα κατάφεραν και φυσικά η Ευρώπη έχει περάσει από πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις και κατάφερε και συνήλθε. Πρέπει λοιπόν να εξυγχρονίσουμε ε, και να βελτιώσουμε την Ευρώπη σήμερα. Έτσι ώστε η κληρονομιά των πατέρων της Ευρώπης να μην χαθεί στα βιβλία της ιστορίας. Αυτή είναι η Ευρώπη την οποία θέλουμε και είμαστε συλλογικά υπεύθυνοι για αυτήν. Είναι δύσκολη αυτή η προσπάθεια, αλλά ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα αποδείξουμε ότι είμαστε ικανοί. Ας καταστήσουμε τους πατέρες μας περήφανος, ας καταστήσουμε τα παιδιά μας περήφανα και ας επιτρέψουμε στην Ευρώπη να στοχεύσει και να επιστρέψει σε ένα λαμπρότερο μέλλον.